Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar la reunión de la Comisión de Pesca del día de hoy. Καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσουμε με τη συνεδρίαση της Επιτροπής Αλίας. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω. Ξεκινάμε με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης και έχουμε κάποιες αλλαγές, τις οποίες θα ήθελα για τις οποίες θα ήθελα να σας πληροφορήσω. Τα έχουμε πει και με τις πολιτικές ομάδες, αλλά ήθελα να σας πω πως τα σημεία 7 και 14 της ημερήσιας διάταξης, δηλαδή είναι η έκθεση Γιώτοβα όπως επίσης και η παρουσίαση από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου των Αγορών Προϊόντων Αλίας και Ιδατοκαλλιέργειας, θα αναβληθούν για μια επόμενη συνεδρία της ομάδας μας. Το ζήτησε η κυρία Ιώτοβα και επίσης ζήτησε κάτι αντίστοιχο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι λοιπόν δεχόμαστε το αίτημα αυτό. Για τα σημεία 7 και 14 επαναλαμβάνω. Δεύτερον, έχουμε το σημείο 12 που είναι η πράσινη βίβλος από τις προκλήσεις της ευκαιρίες προς ένα κοινό πλαίσιο στρατηγικής για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τον κύριο Βαλέσα, ο οποίος είχε σκοπό να συζητηθεί αύριο στις 25 Τετάρτη το θέμα του. Ε, θα χρειαστεί βέβαια να αναβληθεί γιατί δεν μπορέσαμε να βρούμε τον κύριο Βαλέσα και να καταφέρουμε να έρθει στην αυριανή πρωινή μας συνεδρίαση. Για το σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης, όπως σας είπα, ε, δεν θα συζητηθεί. Έχουμε το 8, το οποίο έχουμε προβλέψει για τις 4.30 και κλεισμένων των θυρών. Μόλις τελειώσουμε λοιπόν με το σημείο 6, δηλαδή μάλλον στις 4 παρατέταρτο θα το συζητήσουμε. Άρα λοιπόν να έχετε υπόψη ότι θα συζητηθεί όχι στις 4.30 αλλά νωρίτερα. Έχουμε επίσης και τα διάφορα τα οποία βρίσκεται... Α, και θα ήθελα επίσης να σας υπενθυμίσω ότι η σημερινή συζήτηση βγαίνει απευθείας ε, μεταδίδεται απευθεία από την πύλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λοιπόν, με αυτέ τι μικρέ αλλαγέ εγκρίνει τη μερίσια διάταξη τη σημερινή συνεδρίαση. Έχουμε επίση ω δεύτερο σημείο την έγκριση των πρακτικών τη συνεδρίασης τη 4 η Απριλίου και τη 12 η και 13 η Απριλίου τρέχοντο. Εάν λοιπόν σήμερα ή αύριο δεν ακουστούν ή δεν υποβληθούν αντιρρήσει, θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται τα πρακτικά. Ανακοινώσει τη Προέδρου. Στο σημείο αυτό δεν έχω τίποτα να πω. Μπορώ να περάσω λοιπόν στις ψηφοφορίες. Καταρχήν έχουμε την πρώτη ψηφοφορία για τη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Σαοτομέ και Πρίνσιπε. Ο κύριος Καπούλα Σάντος είναι ο εισηγητής στην περίπτωση αυτή, ο οποίος μου είπε πως γίνεται παράλληλα και στην Επιτροπή Γεωργίας μια ψηφοφορία για ένα θέμα για το οποίο επίση ήταν εισηγητή και επειδή υπάρχει αυτή η χρονική σύμπτωση δεν έχει τη δυνατότητα να παραστεί σήμερα. Μα είπε όμως πως μπορεί να υποβληθεί η έκθεση αυτή για ψηφοφορία. Δεν έχει κανένα σημείο το οποίο να είναι σε κρεμότητα. Έχει συζητηθεί αρκετέ φορέ στην ομάδα μα. Την γνωρίζετε την έκθεση αυτή. Ξέρετε τι έχουν πει οι γνωμοδοτήσεις των Επιτροπών Ανάπτυξης και προπολογισμού ΔΕΒΕ και Budget, άρα λοιπόν μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Ωραία λοιπόν. 118 γάμα της ε, συνθήκης, ε, έγκριση του σχεδίου έκθεσης Έχετε όλοι μαζί την κάρτα και την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ωραία, θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Η πρόταση για το καθορισμό των αλληλευτικών δυνατοτήτων, συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Κοινότητα, Λαϊκή Δημοκρατία, Άτομα και Πρίνσιπε, εισηγητή ο κύριο Καπούλα Σάντο. Είμαστε έτοιμοι. Θέλετε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ωραία λοιπόν, κλείνει η ψηφοφορία. Τι μου ζητήσατε να γίνει κλειστή ψηφοφορία. 19 υπέρ, 17 κατά, μία αποχή, άρα λοιπόν εγκρίνεται με την ηλεκτρονική ψηφοφορία, μέσω της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας συγχαίρουμε τον κύριο Καπούλα Σάντος και μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Να σας πω βέβαια πως την Ολομέλεια ε, του Ιουνίου θα ε, ψηφιστεί και αυτή η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και των Σεχελών. Είναι το δεύτερο σημείο, έχει συζητηθεί αρκετές φορές στην ομάδα μας. Έχουμε την έκθεση του κυρίου Καντέ, έχουμε τις γνωμοδοτήσεις από τις Επιτροπές Ανάπτυξης και Προϋπολογισμού. Μπορούμε λοιπόν να ακολουθήσουμε τη συνήθεια διαδικασία με έκριση σχεδίου έκθεσης. Αν δεν θέλει κανείς να λάβει το λόγο, ξεκινάει η ψηφοφορία για αυτό το νέο πρωτόκολλο. Ξεκινάει Ξεκινάει λοιπόν η ψηφοφορία αυτή τη στιγμή ηλεκτρονικά. Λίγη ψηφοφορία. Και αυτή εγκρίνεται 19 υπέρ, 17 κατά ε, και έχουμε και ε, ε, δεν έχουμε καμία αποχή. Περνάει και αυτή λοιπόν στην Ολομέλεια του Ιουνίου. Νομίζω ότι χρειάζεται να χειροκροτήσουμε ε, τους συναδέλφους. Περνάμε στο σημείο 6 που είναι η γνωμοδότηση Λόβεν για την καταπολέμηση της παράνομης αλληλείας σε παγκόσμιο επίπεδο και ποιος θα είναι ο ρόλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρία λοιπόν ε, Λοβά, έχετε προετοιμάσει αυτή την έκθεση. Οι, επιτροπές, ε, οι επιτροπές ε, περιβάλλοντος και ανάπτυξης έχουν γνωμοδοτήσει. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Λοβέν και μετά θα προχωρήσουμε στην ανταλλαγή απόψεων. Η εισηγήτρια λοιπόν έχει το λόγο. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Όπως είπε και η Πρόεδρος, αυτό είναι το σχέδιο έκθεσης. Μετά βέβαια και τα δύο έγγραφα εργασίας. Μία για για τα πόδα και άλλο ένα για τα διεθνή βήματα τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν στην καταπολέμηση της ε, λαθραλίας σε διεθνή ύδατα. Εδώ λοιπόν έχουμε επιτέλους αυτή, αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης και θα ήθελα να σας εξηγήσω ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα. Να σας πω ότι η λαθραλία, η αλληλεία η οποία δεν δηλώνεται, καλύπτει το 15% του παγκόσμιου αλληλεύματος. Και αυτά βέβαια πρόκειται για απλούς υπολογισμούς, γιατί είναι πολύ δύσκολο να ε, βρει κανείς ποια είναι τα ακριβά, ακριβή στοιχεία. Μιλάμε όμως για κάτι μεταξύ 11 και 26 εκατομμυρίων τόνων ετησίως. Ε, είναι ε, αποτέλεσμα λαθραλίας. Τι σημαίνει αυτό. πως η Λαθραλία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγός αλλιευμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό όχι μόνο διακινδυνεύει την βιωσιμότητα των αλλιευμάτων, ε, δημιουργεί προβλήματα για τη βιοπικιλότητα και την επιβίωση αυτής και πάρα πολλά από αυτά τα θέματα τα έχω τοποθετήσει ε, στην ε, γνωμοδότηση μου το 72% του πλανήτη είναι ωκεανή, αλλά το 90% της βιόσφαιρας του πλανήτη μας είναι ωκεανή, οι θάλασσες. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι πάνω από δύο τρίτα αυτή τη ε, βιόσφαιρας βρίσκεται σε διεθνή ύδατα εκτός εθνικής δικαιοδοσία. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε το εργαλείο των διεθνών συμφωνιών και βέβαια πρέπει να καταβάλουμε και κάποιες διεθνείς προσπάθειες, προσπάθειε σε διεθνή επίπεδα έτσι ώστε να πατάξουμε αυτή την ανεξέλεγκτη άντληση των, του φυσικού αυτού πόρου από τα παγκοσμία ύδατα. Ένα άλλο σημείο το οποίο τονίζω εδώ είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζουμε πως εμείς έχουμε αναλάβει στην Αγκόγια τη σχετική δέσμευση έτσι ώστε να φρενάρουμε την μείωση της ε, βιοπικιλότητας, αλλά στα πλαίσια της ατζέντα για το 2020 οι επιδόσεις μας είναι μάλλον μέτριες, γιατί είχαμε ε, αναλάβει κάποιες ε, δεσμεύσεις για μείωση αυτής της παράνομη αλίας μέχρι το 2010. Δεν πετύχαμε εκεί του στόχου μας. Άρα λοιπόν το πιο προφανές βήμα είναι αυτή, αυτό το είδο αλίας να περιοριστεί. Είμαστε από του βασικούς παίκτε ε, στο χώρο αυτό, γιατί είμαστε και μεγάλος εισαγωγέας αλλιευμάτων, αλλά και έχουμε μεγάλη αλλιευτική βιομηχανία. Είμαστε λοιπόν η μεγαλύτερη αγορά ε, για αυτά τα προϊόντα και μπορούμε πολλά να κάνουμε, όχι μόνο με την ιδιότητα ε, της μεγάλης πολιτικής δύναμης στην παγκόσμια σκηνή, αλλά γιατί εκπροσωπούμε και μεγάλα εμπορικά συμφέροντα και μπορούμε να κάνουμε και πολλά μέσω εισαγωγικών ε, πολιτικών που θα ακολουθήσουμε. Θα ήθελα καταρχήν εδώ να τονίσουμε το ποιος θα είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα πρέπει να είναι υποδειγματική στις δράσεις της, Έχουμε και τον σχετικό κανονισμό που ετεθηκε για από 1η ε, Ιανουαρίου τρέχοντος, που αποτελεί βασικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Και νομίζω πως είναι ένα εξαιρετικό πρώτο βήμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα κράτη-μέλη να έχουν αρκετούς πόρους στη διάθεσή τους και ανθρώπινους και οικονομικούς, αλλά να έχουν και τις τεχνολογικές ε, δυνατότητες που χρειάζονται για να εφαρμόσουν τον κανονισμό αυτό και να μην αποφύγουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις και πρόστιμο όταν αυτό χρειάζεται, γιατί βεβαίως εδώ διακυβεύεται και η ίδια αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επίσης ανταλλαγή πληροφοριών για τις αλληλευτικές δραστηριότητες, για την λαθραλία, για την παράνομη αλληλεία μεταξύ με κρατών μελών, με την Κομισιόν και με τον φορέα που επιβλέπει είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θεωρούμε ότι χρειάζεται μία ετήσια παρακολούθηση των επιδόσεων των κρατών μελών σε επίπεδο εφαρμογή της αλληλευτικής πολιτικής και κυρίως εφαρμογής των ευρω των πολιτικών και των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντική και θα πρέπει να δημοσιεύονται αυτοί οι κατάλογοι επιδόσεων και να δημοσιοποιούνται έτσι ώστε σε κάθε επίπεδο ε, να στηρίξουμε και τα αναπτυσσόμενα κράτη έτσι ώστε τους κανονισμούς αυτούς να τους εφαρμόσουν και αυτά με συνοδευτικά έγγραφα για τα λιεύματα τα οποία θα είναι αξιόπιστα, όπως επίσης και με ενίσχυση των εθνικών τους δυνατοτήτων για έλεγχο και υποπτία και παρακολούθηση. Για τους λιμένες δε, πιστεύω ότι για την εκφόρτωση στις χώρες αυτές και εκεί θα πρέπει να καταβάλουμε τις σχετικές προσπάθειες. Έχουμε ακούσει πολλές προτάσεις, πολλές έχουμε συμπεριλάβει στην έκθεσή μας. Για παράδειγμα, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις διάφορες διεθνείς ε, συμφωνίες, για παράδειγμα, για τη Συμφωνία για την εκφόρτωση στους λιμένες εκφόρτωση, την συμμόρφωση με τους κανονισμούς του ΟΗΕ για την αερία, να τα θέτει ως προϋποθέσεις για να συμμετέχουν τα διάφορα κράτη στο Γενικό Σύστημα Προτιμήσεων γιατί αυτό θα αποτελούσε και ένα πολύ θετικό βήμα για τα αναπτυσσόμενα κράτη. Δηλαδή το να καταφέρουν να ξεπεράσουν αυτή την πληγή που είναι η λαθραλία στα διεθνή ύδατα, κοντά στα εθνικά ύδατα των χωρών αυτών. Γιατί ξέρετε ότι η απώλεια εισοδήματο για τα κράτη θα είναι πολύ σημαντική από αυτήν την λαθραλία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενισχύσει και τις οργανώσεις περιφερειακές αλίας και τα περιφερειακά γραφεία, ε, να δουν με τι γίνεται με τις επιτροπές συμμόρφωσης και πώς μπορεί να ενισχυθεί ο ρόλος τους έτσι ώστε τα συμβαλόμενα μέρη να ελέγχονται. Και όπου βέβαια είναι απαραίτητο θα πρέπει να επιβάλλονται ε, και αποτρεπτικές κυρώσεις. Χρειαζόμαστε μητρώα αλληλευτικών σκαφών σε όλες τις περιφερειακές ε, σε επιφυριακά βήματα. Και θα πρέπει να δούμε και τι θα γίνει με το μαύρο κατάλογο σκαφών ε, που έχουν ε, βρεθεί να λαθραλιεύουν. Δεν μου αρέσει η έννοια του λευκού καταλόγου, δηλαδή τα σκάφτα που επιτρέπεται να αλλιεύουν, αλλά τουλάχιστον όσους έχουμε ε, όσοι έχουν καταγγελθεί και βρεθεί με παράνομα αλλιεύματα θα πρέπει να υποστούν κάποιες κυρώσεις και ενδεχομένως να τοποθετηθούν σε μαύρη λίστα. Κάτι ακόμα που χρειαζόμαστε είναι αυτές οι συμφωνίες να επεκταθούν, να δούμε ποια είναι η εντολή, ε, ποια είναι η γεωγραφική περιοχή που καλύπτουν, να καλύπτονται όλα τα είδη ή τουλάχιστον όλα τα είδη αλλιευμάτων στα διεθνή ύδατα. Αυτή τη στιγμή μόνο ένα τμήμα των ειδών αυτή τη στιγμή είναι υποκείμενο αντικείμενο διαχείρισης από αυτούς τους περιφερειακούς οργανισμούς αλίας. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πως έχουμε αναλάβει μια δέσμευση να φρενάρουμε την μείωση της βιοπικιλότητας και το μόνο εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή σε επίπεδο διεθνού κοινότητα είναι αυτό το οποίο παρουσιάζει αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον όσον αφορά την αλληλεία εκτός χωρικών υδάτων, εθνικών χωρικών υδάτων. Γιατί πρέπει να εξασφαλίσουμε στις επόμενες γενιές πως τα διάφορα είδη θα διατηρηθούν και πως η βιοποιλικιλότητα στα διεθνή ύδατα δεν θα καταστραφεί με την ταχύτητα που καταστρέφεται σήμερα. Θα πρέπει λοιπόν η εντολή να επεκταθεί ε, και αυτό είναι, κάτι, αυτό το Περιφερειακό Συμβουλίο και αυτό το έχουμε προτείνει. Βεβαίως και στηρίζουμε την πρωτοβουλία του ΦΑΟ για να έχουμε ένα παγκόσμιο μητρό αλληλευτικών σκαφών, το οποίο θα είναι υποχρεωτικό και θα είναι όλα τα σκάφη πάνω από 18 που θα εντάσσονται σε αυτόν. Θα πρέπει να γίνει βέβαια και κάποια ε, και κάποια αξιολόγηση των διαφόρων κρατών και των επιδόσεων των ε, κρατών σημαία, έτσι ώστε να πιέζονται τα κράτη τα οποία δεν συμμορφώνονται ή δεν σέβονται τι διεθνεί υποχρεώσει του. Θέλουμε να δημιουργηθεί ένα νέο σώμα, ένας νέος φορέας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ έτσι ώστε να ελέγχει και τα κράτη σημαία αλλά και ε, τα περιφερειακά αυτά ε, συμβούλια και τα περιφερειακά προγράμματα παρατήρησης, τα πόδα. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει την πρωτοβουλία να συνεργαστεί με τις χώρες οι οποίες είναι οι βασικές αγορές για τα λιεύματα, Κίνα, Ιαπωνία, ΙΠΑ για παράδειγμα, έτσι ώστε να βρούμε ένα κοινό τόπο για να έχουμε τα απαραίτητα νομικά εργαλεία που θα επιτρέψουν να πατάξουμε την εμπορία λαθραλιευμάτων. Αυτό το οποίο μας ενθαρρύνει ιδιαίτερα είναι μια δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λέει πως χρειάζεται ε, να προωθήσουμε ένα καθεστώς ε, ένα παγκόσμιο καθεστώς πιστοποίησης αλλιεύματος, κάτι τέτοιο θα ήταν ιδιαίτερα παρήγορο. Επίσης, έχουμε το θέμα ε, του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος στα πλαίσια αυτής της παράνομης αλλίας και πρόσφατα δημοσιεύθηκε από το Διεθνές Γραφείο ε, για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα των Ηνωμένων Εθνών μια έκθεση για τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι εγκληματικές συμμορίες επεκτείνουν τα συμφέροντά τους για να καλύψουν και τον κλάδο της αλληλείας. Εδώ συμπεριλαμβάνουμε πολύ ανησυχητικά και δυσάρεστα φαινόμενα Έχουμε λοιπόν εδώ την διαφορά, διαφθορά, την ε, σωματεμπορία, την τελωνιακή, ε, ε, τις τελωνιακές παραβάσεις, το έγκλημα. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως δεν είναι μόνο οι κανόνες ε, της περιοντολογικής διατήρησης των ειδών οι οποίοι καταπατώνται και παραβιάζονται εδώ, αλλά και η νομοθεσία ε, στους προηγούμενους κλάδους που σας ανέφερα. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να τονιστεί παραπάνω. Να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι διαστάσεις και πού φτάνει ε, αυτό το έγκλημα και να δούμε πώς μπορούμε χρησιμοποιώντας τα διάφορα, τις διάφορες διεθνείς συμφωνίες να πατάξουμε αυτού του είδους την λαθραλία. Δηλαδή έχουμε την σύμβαση του ΟΗΕ που έχει επικυρωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό ε, για την πάταξη του εγκλήματος και που υποχρεώνονται τα συμβαλόμενα μέρη να συνεργάζονται σε επίπεδο, κατα... σε επίπεδο δίωξης και δικαστικής αρρωγής. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαμε να καταπολεμήσουμε την λαθραλία. Η Ίντερπολ αυτή τη στιγμή ως μία από τις ε, περιοχές ε, προτεραιότητας έχει τοποθετήσει το περιβαλλοντολογικό έγκλημα και θεωρούμε πως η Ίντερπολ θα μπορούσε να αποτελέσει τον κατάλληλο τόπο για συνεργασία, ένα βήμα το οποίο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη στιγμή που διεξάγουμε έρευνες σε θέματα που άπτονται της διεθνούς λαθρελίας. 64% των ωκεανών των διεθνών θαλασσών βρίσκονται εκτός εθνικής κυριαρχίας. Είναι λοιπόν επίγον να φέρουμε σε πέρας κάποιες προσπάθειες για αυτή την ταχύτατη και καταστροφική απώλεια βιοπικιλότητας, όπως επίσης και για την φθορά ε, των ε, θαλασσίων οικοσυστημάτων. Θα πρέπει όλα αυτά ε, να αποτελέσουν προτεραιότητα στο επόμενο, στην, επόμενο, στην επόμενη σύνοδο διάσκεψη για το βιώσιμο περιβάλλον που θα γίνει του χρόνου που βεβαίως θα εορτάσει και την 30 επέτειο του δικαίου της θάλασσας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Ένα, αυτό, λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα πρέπει εκεί να συζητηθούν και κυρίως η διάσταση αυτή των ωκεανών. Ελπίζω λοιπόν με τα σχόλια που θα κάνετε να συνεισφέρετε και εσείς στην συζήτηση αυτής της έκθεσης. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής, η κυρία, ο κύριος Αρσένης. Thank you very much, Madam President. Ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια για την εξαιρετική δουλειά. Προσωπικά προσυπογράφω τα σημεία της έκθεσης. Αλήθεια είναι ότι η Ελία Πλά δεν απειλεί μόνο τη βιοποικιλότητα και τα λιεύματα και τους αλείς σε τελευταία ανάλυση αλλά συνδέεται και με εγκληματικές δραστηριότητες. Με το οργανωμένο έγκλημα, με πολλούς τρόπους συνδέεται. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πολλοί κανονισμοί και πρέπει να εστιάσουμε στη συμμόρφωση. Ήρθε η ώρα λοιπόν να προχωρήσουμε στην εφαρμογή. Ο ρόλος των πόδα είναι πάρα πολύ σημαντικός, είναι κρίσιμη σημασία των πόδα περιφερειακών οργανώσεων ε, διαχείρισης της αλίας και πρέπει να έχουμε τήσια ή περιοδική τέλο πάντων ε, εξέταση και παρακολούθηση των επιδόσεών τους και όταν βλέπουμε κενά στη λειτουργία θέματα που χρήζουν βελτιώσεων όλα αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οπωσδήποτε ως συστάσεις και υποστηρίζω και τη γνώμη της εισηγήτριας ε, σχετικά με τις πρωτοβουλίες του ΦΑΟ ο οποίος έχει αρχίσει πολλές πρωτοβουλίες που τρέχουν ακόμα και είναι αποτελεσματικές από ό,τι φαίνεται στην αντιμετώπιση της παράνομης λαθρέας άναρχης αλίας. Ο κύριος ε, Κούσταυσεν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την Ιζαμπέλα για την πολύ καλή της έκθεση. Αποτελεί μια πολύ καλή βάση Έχουμε ήδη δύο έγγραφα εργασία και ξέρουμε πλέον και φαίνουμε, βλέπουμε περί πρόκειται και πώ μπορούμε να καταπολεμήσουμε αυτό το πρόβλημα. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτούς που κάνουν απάτες. Έχουμε να κάνουμε με την βιωσιμότητα αυτού του χώρου είναι σημαντικό για το περιβάλλον μας, για το οικοσύστημά μας, για τα αποθέματα των αλλιευμάτων, για όλες αυτές τις ψυχές. Και η κυρία Λέβιν, κατά με, θα έπρεπε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στο γεγονός ότι όλα αυτά είναι σημαντικά για τους αλληλείς, για τους έντιμους αλληλείς. Αυτό θα πρέπει να το θίξουμε στην έκθεση, διότι αυτοί που κάνουν απάτες ε, ε, ε, κάνουν ενέργειες που ενδεχομένω σε βάρος των εντύμων λευμάτων. Θα, δώσω, λοιπόν, θα κάποιες τροπολογίες με αυτήν εδώ την οπτική γωνία. Και όπως ελέγχθη λοιπόν είναι γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει ένα σημαντικό ρόλο όσον αφορά τη εισαγωγή προϊόντων αλλιεύσεως. Και θα πρέπει και ο καταναλωτής να καταλαβαίνει να είναι να έχει γνώση του τι ακριβώς αγοράζει. Να ξέρει δηλαδή αν κάτι αγοράζει το οποίο έχει γίνει νομίμως ή όχι. Αυτοί που αγοράζουν λαπίν ε, ε, ψάρι θα πρέπει να ξέρουν αν αυτό που αγοράζουν έχει αλληλευθεί νόμιμα ή όχι. Θα πρέπει δηλαδή να κάνουν κάποιες ενέργειες ώστε να ανοιχνευθεί όλη η οχι θα πρεπει δηλαδη να κανω καποιες ενεργειες ωστε να ανοιχνευθει ολη η διαδικασια του προϊόντος και πώς αυτό καταλήγει στον ε, καταναλωτή για να προστατευθεί ο καταναλωτής έναντι των παρανόμων Φέρει Φερρυπίν ε, όταν αγοράζει κανείς ε, σιγάρα γίνεται ένα του τόσο να μην αγοράζει κανείς σιγάρα τα οποία είναι, έχουν εισαχθεί παράνομα. Αυτό θα πρέπει να ισχύει και για τα λεύματα. Στην Ευρώπη λοιπόν θα πρέπει να βάλουμε μια τάξη τάξη στα του οίκου μα καταρχήν, όχι μόνο αυτά, αυτά που γίνονται έξω. Θα πρέπει να δώσουμε μια έμφαση, να λάβουμε μέτρα τα οποία να ισχύουν εδώ σε εμά. Περιμένω λοιπόν να την περαιτέρω συνέχεια τη εκθέσεω αυτή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ριβελίνη. Naturalmente mi congratulo e mi complimento. Μα φυσικά. Συγχαίρω την εισηγήτριά μας να μην επαναλάβω για τις αρνητικές επιπτώσεις της παράνομης αλίας που είναι, αποτελούν και, μια, και ένα θέμητο ανταγωνισμό και αποβαίνουν και εις βάρος του περιβάλλοντος. Εγώ να επενθυμίσω τα ότι η διάσκεψη ΦΑΟ ε, αρχές της χρονιάς έχει καταλήξει σε ένα νέο σύστημα ε, σήμανσης για να μπορέσει κανείς να καταπολεμήσει την παράνομη αλία. Έχουν συζητηθεί κάποιοι κανόνες στα πλαίσια του ΦΑΟ και αυτοί οι κανόνες θα πρέπει να αναφερθούν ρητά στην έκθεση της κυρίας Λέβιν αναφέροντας φυσικά το νέο σύστημα σήμανσης που είναι πολύ συγκεκριμένο ποια είναι η ζώνη στην οποία φέρει το έχει γίνει η αλίευση, ποια είναι τα είδη, και όλα αυτά τα στοιχεία είναι σημαντικά. Να το λάβει λοιπόν αυτό υπόψη η κυρία Λέβιν. Τώρα, κάποιες άλλες παρατηρήσεις. Για το δεύτερο μέρος της εκθέσεως, Λέβιν. Η ενέσχυση των ελέγχων ε, στις, ε, εκτός ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ξέρουμε για τις διαδικασίες εκεί που υπάρχουν με έναν τρόπο θα λέγαμε μη νόμιμο, κλείνει κανείς τα μάτια και διακινούνται αλλιεύματα τα οποία έχουν αλλιευθεί παρανόμως. Άρα θέλουμε μια ενίσχυση σε διεθνές επίπεδο για έλεγχο, συνεργασία φυσικά ανάμεσα σε χώρες, σε χώρες ούτως ώστε <coughs> συγγνώμη, να υπάρξει ε, ένας έλεγχος, έλεγχος των ποσοστώσεων και να υπάρχει ένα συλλογικό έλεγχος τελικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να θέσει εφαρμογή ένα τέτοιο σύστημα καταρχήν για να για να πατάξει την παράνομη αλληλεία και φυσικά για να δώσει και το καλό παράδειγμα στις τρίτες χώρες, στις στοχές χώρες Φερρυπίν της Αφρικής που πλήττονται από την παράνομη αλληλεία. Τον Ιούνιο θα γίνει μια συνάντηση σε σχέση με αυτό, με βάση την ιδέα της δημιουργίας ε, ε, μιας υπηρεσίας ακτοφυλακής ευρωπαϊ... ευρωπαϊκής και φυσικά όλοι είναι πρόσθετοι να συμβάλλουν σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ την εισηγήτρια και να της πω ότι είναι εξαιρετική η μορφή που έχει αυτή η έκθεση. Πιστεύω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ότι μπορεί, απλώς πρέπει, πρέπει να αποτελέσει το κομβικό σημείο για, την, για τον έλεγχο της λαθραλίας. Γιατί έχουμε πολλούς αλληλείς, γιατί είμαστε μεγάλο, μεγάλη εισαγωγική αγορά και γιατί έχουμε υπογράψει πολλές διεθνείς συνθήκες που μπορούν να γύρουν την πλάστικα υπέρ μας αυτή τη μάχη κατά της λαθραλίας θα πρέπει μέσω των εμπορικών μας πολιτικών να τοποθετήσουμε και αυτή τη διάσταση, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε την αθρελία. Επίσης, θα πρέπει να δούμε ε, πώς μπορούμε να δημοσιοποιούμε τις επιδόσεις όλων. Αυτό που χρειάζεται όμως τα στοιχεία αυτά και τα κριτήρια αξιολόγηση να χρησιμοποιούνται με πανομοιότυπο τρόπο έτσι ώστε να βαθμολογούνται όλοι σύμφωνα με την ίδια κλίμακα. Αυτό που είναι σημαντικό είναι η εκφόρτωση των οπών αλλά επίσης και των κοντέινερ γιατί ο έλεγχος αυτός είναι πολύ σημαντικός. Έτσι μπορούμε να εξασφαλίσουμε και την επιστημιστική ασφάλεια μέσω της ιχνηλασιμότητας. Εμείς έχουμε τροπολογίες τις οποίες πιστεύουμε πως θα βελτιώσουν το κείμενο, θα μιλήσουμε με την εισηγήτρια και θα συνεργαστούμε μαζί της γιατί συμφωνούμε απόλυτα πως τέτοιου είδους εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις μας βοηθούν στην προσπάθεια που κάνουμε για να περιορίσουμε τη λαθραλία. Σας ευχαριστώ πολύ ο κύριος Κέλλη, ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν να ευχαριστήσω την Ζαμπέλα για το έργο της, για την έκθεσή της. Είναι γεγονό ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της παράνομης αλληλείας είναι πολύ σημαντικός. Υπάρχουν οι που έχουν να κάνουν με την υγεία, την ε, ε, σωστή αλλίευση και το περιβάλλον. Προτείνω, λοιπόν κάποιες λύσεις για να καταπολεμηθεί αυτό το, ε, το πρόβλημα και φυσικά για να προστατευτεί και η ευρωπαϊκή παραγωγή. Αλλά φυσικά πρέπει οι χώρες μέλη και οι οργανισμοί, οι διεθνείς, οι οποίοι θα πρέπει να συνεργαστούν, σημαντικό να το πούμε, ούτω ώστε να εξαλειφθεί αυτό το πρόβλημα της παράνομης αλίας. Όπως και να το κάνουμε, συμφωνώ ότι για το θέμα τη, του συστήματο γενικευμένων προτιμήσεων και είναι ένα σημαντικό θέμα αυτό. Ε, βλέπει κανείς ότι σε ορισμένε χώρες, με τι οποίε έχουμε συμφωνίε. κυρίως χώρες ε, οι οποίες, ε, τις οποίες πραγματικά γίνεται συστηματική παράνομη αλία. Τα προϊόντα αυτά δεν θα πρέπει να μπαίνουν στην ε, ευρωπαϊκή επικράτεια, εισάγονται εδώ και γι' αυτό χρειάζεται ένας σύστημα ελέγχου φυσικά. Όλα αυτά πηγαίνουν προς σωστή κατεύθυνση. Και βλέπουμε το παράδειγμα που ανέφερε πριν από λίγο για τις ασιατικές χώρες, όπου πραγματικά εξαντλούνται τα αποθέματα, δεν γίνεται σεβασμό στο διεθνού δικαίου, γι' αυτό θα πρέπει να σταματήσει αυτό. Και είναι και αυτό μέρος του αγώνα που γίνεται κατά της παράνομης αλίας. Διαπιστώνω ότι αυτό το θέμα ξεπερνάει τα θέματα που έχουν να κάνουν μόνο με την αλία, όπως είπαν και ορισμένοι συνάδελφοι, αγγίζουμε πλέον και θέματα οργανωμένου εγκλήματο. Έχουμε να κάνουμε το σεβασμό του δικαιώματο στην και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε τελική ανάλυση. Αν υπάρχει ένα θέμα στο οποίο όλοι συμφωνούμε, ε, ειλικρινά, ε, είναι αυτό εδώ όπου θέλουμε να καταπολεμήσουμε την παράνομη αλία και θα υποστήριξουμε όντως την έκθεση της Ιζαμπέλας Λεβίν. Ο κύριος Μπέμπης. Ευχαριστώ. Χαιρετίζω την ομοφωνία στην Επιτροπή υπέρ της ανάληψης δράσης κατά της παράνομης αλίας. Δύο ερωτήσεις προς την εισηγήτρια την Κομισιόν. Η εισηγήτρια υπογραμμίζει τη σημασία της πολιτικής βούλησης των κυβερνήσεων που πρέπει να αναλάβουν δράση για την αντιμετώπιση του προβλήματος στο έδαφος τους και κάνει προτάσεις ε, ε, να κατονομάζονται οι υπεύθυνοι και έτσι να ντροπιάζονται όταν δεν αναλαμβάνουν δράση. Πώς θα μετρήσουμε όμως τις επιδόσεις, ε, δηλαδή Παγκοσμίω εικασίε υπάρχουν μόνο για την παράνομη αλία και την έκταση που έχει. Είναι πολύ δύσκολο να είναι ακριβή τα στοιχεία. Καμιά φορά όμως η ποσότητα της παράνομης αλίας ε, δεν μπορεί να μετρηθεί επακριβώ. Εικάζουμε μόνο, οπότε πώ θα μετρήσετε και την πολιτική βούληση των κρατών μελών να την καταπολεμήσουν. Δεύτερη ερώτηση. Ε, το αίτημα σχετικά με την ε, καταχώρηση του Μητρώου όλων των αλλιευτικών σκαφών και δημοσίευση των δεδομένων. Τα αλλιεύματα, τα ψάρια είναι δημόσιο αγαθό. Η κοινή γνώμη έχει δικαίωμα να γνωρίζει ποιος αλλιεύει αυτό το δημόσιο αγαθό. Τον πόρο πρέπει λοιπόν να είναι κοινέ πληροφορίες και ε, έχει να κάνει και με τα μεταβιβάσιμα δικαιώματα και όλα αυτά. Η αρχή αυτή έτσι γίνεται ακόμα πιο αυστηρή και ισχυρή. Τα έχουν περάσει όμω πολλά χρόνια απραξία. Ποιο είναι ο λόγο, γιατί μέχρι τώρα δεν κάναμε τίποτε. Κυρία Πέτρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια για την εργασία της αυτή, η οποία υποστηρίζεται γενικότερα από εμάς ε, είναι πολύ σημαντικό θέμα. Τα ψάρια συμφωνούμε πάνω σε αυτό. Θα προσθέσω εδώ όμως ότι αυτό που θα ήθελα να πω δεν έχει παρουσιαστεί έτσι τόσο ξεκάθαρα όσο θα ήθελα. Ω συμβολή μου προς την έκθεση, βέβαια είναι ολοκληρωμένη η έκθεση, αλλά μπορούμε παρόλα αυτά να προσθέσουμε κάποια θέματα εκτός από αυτά που έχουν αναφερθεί για την καταπολέμηση της παράνομης αλίας. Πιστεύουμε ότι θα επιτύχουμε στην καταπολέμηση της παράνομης αλίας αν λάβουμε υπόψη μας όλες τις πτυχές με τρόπο συνεπή. Η λύση πρέπει να είναι συνεπής, συνεκτική. Και σε αυτά τα πλαίσια θέλω να τονίσω τη σημασία ενός νέου κανονιστικού πλαισίου που ελπίζουμε να προκύψει σύντομα, ίσως τον Ιούνιο. Πρέπει να είναι αποτελεσματικό για να καταπολεμήσει την παράνομη αλληλεία. Ένα θέμα είναι τα δικά μας μοντέλα διαχείρισης. Υπάρχουν καμιά φορά νομικοί περιορισμοί που δεν συνάδουν με την κατάσταση των αποθεμάτων, των νύχθη αποθεμάτων. Και έτσι μεταξύ των αλλιέων δημιουργείται η επιθυμία να συνεχίσουν τις πρακτικές τους παρόλο που αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι προς όφελός τους αυτό. Κάτι άλλο επίσης που θέλω να πω, πέρα από την καταπολέμηση της παράνομης ε, αλληλείας, Ιδιαίτερα στα είδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι νομίζω σημαντικό να συσταθούν μηχανισμοί ώστε ο οπορτουνισμός, η ευκαιριακή προσέγγιση να καταπολεμηθεί ο σύμμαχος της παράνομης αλίας. Θα πρέπει να έχουμε τις προϋποθέσεις εκείνες ώστε ο κόσμος που δραστηριοποιείται στον τομέα να κατανοήσει ότι να κερδίσει μόνο έχει αν εγκαταλείψει αυτές τις παράνομες πρακτικές. Πρέπει να αποκτήσουν εκείνη υπευθυνότητα και θα πρέπει και εκείνοι να συμμετέχουν στην καταπολέμηση της παράνομης αλίας. Έτσι θα υπάρχουν ωφέλη για όλους. Αυτά είναι κάποιες παρατηρήσεις που νομίζω ότι καλό θα ήταν να γίνουν για να συμβάλλω κι εγώ στην πάρα πολύ αξιόλογη έκθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν κάποια σημεία με τα οποία θα συμφωνήσω ιδιαίτερα στην έκθεση και θα τις απευθύνω και κάποιες ερωτήσεις κυρία Λόιβιν. Καταρχήν μίλησε για μια σύνδεση μεταξύ οργανωμένου εγκλήματος και προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε με την αλληλεία. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το υπογραμμίσουμε γιατί ακούμε τα όσα λένε οι αρχές οι οποίες είναι υπεύθυνε για την ασφάλεια στη θάλασσα και στους ωκεανούς ή τα όσα λένε οι αρχές που είναι υπεύθυνε είτε σε περίπτωση πειρατείας είτε ελαθραλίας και βλέπουμε πως υπάρχει ένα έλλειμμα δυνατότητας ελέγχου ε, και εποπτείας σε όλες τις θάλασσες. Νομίζω ότι πολύ σωστά αυτό τονίζεται στην ε, γνωμοδότηση. Το πρόβλημα είναι τι είδους συστάσεις μπορούμε να προτείνουμε και πώς μπορούν αυτές στην πράξη να εφαρμοστούν. Προλίγου είπε κάποιος συνάδελφος που χρειαζόμαστε ακτοφυλακή. Να σας πω πως στη Γαλλία Έχουμε ένα σύστημα ε, με τους ε, επάρχους που είναι υπεύθυνοι για τη θάλασσα και ρυθμίζουν και το θέμα της θαλάσσιας κυκλοφορίας, ε, ελέγχουν και την αλία και θέματα ασφάλειας που άπτονται αυτής και έτσι υπάρχει αυτή τη στιγμή διοίκηση της ακτοφυλακής πολύ αποτελεσματική. Και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Εγώ πρέπει να σας πω πως στο παρελθόν ασχολήθηκα με το θέμα του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και πήγα και στον ΟΗΕ σε κάποιες ανταλλαγές ε, απόψεων και σε συναντήσεις που ήταν ε, εξαιρετικές. Αλλά τη στιγμή του συντονισμού στην πράξη δεν είμαστε αρκετά αποδοτικοί και θα με συνέχεια σε αυτές τις εξαιρετικές εκθέσεις που προετοιμάζονται. Γι' αυτό λοιπόν ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει ποια είναι τα πρακτικά μέτρα συντονισμού που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην πράξη έτσι ώστε να αξιολογήσουμε σήμερα τα μέσα που έχουν ήδη στα τα κράτη-μέλη στη διάθεσή τους για να συνεργαστούμε, επαναλαμβάνω, στην πράξη ε, στα ύδατα τα οποία είναι υπό την εθνική μας κυριαρχία. Επαναλαμβάνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο άρθρο 14 μιλάμε για ένα νέο φορέα ο οποίος θα μπορούσε να συσταθεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες εκεί, να μας πείτε ακριβώς τι έχει κατά νου. Και να μας πει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς θα αντιμετωπίζει. Και το τρίτο στοιχείο είναι για την θέση σε εμπορία. Πώς μπορούμε εμείς να ξεπεράσουμε το όσα έχουμε στο άρθρο 15, δηλαδή η έννοια της υπευθυνότητας η οποία, την οποία φέρει το κράτος εμπορίας. Δηλαδή έτσι ώστε αυτά τα λαθραλιεύματα να μην μπορούν να μπουν στην αγορά. Νομίζω ότι αυτό ταιριάζει με τα όσα προσπαθεί να κάνει η συγκητριά μας. Ε, τώρα για την ίχνη συλλομότητα και αυτή μας εξασφαλίζει κάποιες δυνατότητες, αλλά νομίζω ότι εδώ πρέπει να πλησιάσουμε την πρόταση αυτή με πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Ο κύριος Μιλάνα. Και εγώ επίσης να χαιρετήσω την Ιζαβέλα για την πολύ καλή της έκθεση που είναι πολύ σημαντική. Η κυρία Τρότμαν έκανε μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση. Υπάρχει παράνομη ελεία που κα... καταλήγει στο νόμιμο εμπόριο και κάποια άλλη που καταλήγει σε ένα παράνομο εμπόριο. Θα πρέπει να τα δούμε αυτά τα. Θα πρέπει να δούμε όλη αυτή τη διαδικασία, όχι μόνο το τι ακριβώ γίνεται στου ωκεανού. Ο ωκεανό δεν έχει όρια. τα δράματα ξεπερνάνε τα όρια αυτά και καταλήγουν στην αγορά. Και γι' αυτό συμφωνώ με την κυρία Τράτμαν με αυτή την παρατήρηση. Τώρα μια άλλη πτυχή που είναι εξίσου σημαντική. Έχει να κάνει με την Ευρώπη μας. Θεωρώ λοιπόν ότι, ότι δεν ασχολούμαστε όσο πρέπει για το θέμα της ε, για το τι το τι ε, ακριβώς γίνεται πέρα από τα όρια την επικράτεια την ευρωπαϊκή. Έχουμε επίσης και ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με την, ε, ε, την αλία σαν χόμπι. Αυτή είναι ένα σημαντικό θέμα, το οποίο συνδέεται με την παράνομη αλληλεία και θα πρέπει να ελεγχθεί. Θεωρώ λοιπόν ότι αν πραγματικά μας είναι προσφυλές αυτό το θέμα της βιοπικιλότητας των ωκεανών κτλ. Θα πρέπει λοιπόν να, δείξουμε, ε, να έχουμε, είμαστε πολύ πιο αυστηροί όσον αφορά τους κανόνες και στην αλία σαν χόμπι. Διότι σε αυτόν εδώ το χώρο πολύ συχνά διαπιστώνει κανείς ότι γίνεται μια ε, γίνεται μέσω δηλαδή αυτού του χώρου μια, ε, ένα πέρασμα παράνομης αλίας. ήτη θα πρέπει να δώσουμε, μια, ε, να δώσουμε έμφαση σε αυτό. Να αναφερθώ τώρα εδώ και στη, στο, στη Μεσόγειο, διότι εδώ πέρα έχουμε με μια μεγάλη δραστηριότητα και υπάρχει και μια σκιά ανάμεσα στις δραστηριότητες που είναι χόμπι ή όχι. Και πρέπει να ξεχωρίσουμε, να κάνουμε μια κατηγοροποίηση του σωστούς ε, και εμείς ε, χόμπι αλίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι όλη η διαδικασία σύνταξης της έκθεσης ήταν πραγματικά άριστη και θα ήθελα να σας συγχαρώ κι εγώ όπως οι συνάδελφοι, αγαπητή Ισαμπέλα. Και χαίρομαι που μπορέσαμε να συνεργαστούμε τόσο στενά στο θέμα αυτό. Την περασμένη εβδομάδα είχα πάει στο Βιετνάμ για να δω τι γίνεται με το θέμα της εμπορίας του Παγκάσιους και πρέπει να σας πω πως εντυπωσιάστηκα στο ποταμό Μεκόγκ. Πήγα και στο Ανόη να συναντηθώ με το Υπουργείο Αλίας και πρέπει να σα πω πω τα θέματα που αντιμετωπίζει εκεί ο υπουργό, εκτό από το γεγονό πω μειώνεται το απόθεμα, είναι η λαθραλία, ανισχούν ιδιαίτερα οι Βιετναμέζοι στο θέμα αυτό, όπως εμείς, το γεγονός πως το 40% του στόλου αυτή τη στιγμή έχει δέσει στα λιμάνια του Βιετνάμ γιατί έχει αυξηθεί το κόστος καυσίμων. Λοιπόν, μην νομίζετε ότι μόνο εμείς έχουμε πληγεί από τα προβλήματα αυτά. Όπου ταξιδέψει κανείς, διαπιστώνει πως όλοι αντιμετωπίζουν τελικά τις ίδιες δυσκολίες. Βέβαια, θα συμφωνήσω με τα όσα είπε και ο κύριος Μιλάνα μόλις. 11 με 26 εκατομμύρια τόνοι, όπως λέει η γνωμοδότηση, είναι λαθραλίευμα. Και όλο αυτό το αλίευμα μπαίνει στην αγορά κάπως. Πάρα πολύ από αυτό στη δική μας αγορά, γιατί εμείς καλύπτουμε μόνο το 60% των δικών μας αναγκών. Άρα λοιπόν λαθρεία ε, στην ε, ευρωπαϊκή αγορά. 40% λοιπόν αυτού του ε, ελλείμματος προκύπτει από την εισαγωγή των ειδών αυτών ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως η μεταφόρτωση αυτών των αλλιευμάτων γίνεται στα διεθνή ύδατα που δεν υπάρχει εθνική δικαιοδοσία και μετά αναμειγνύεται με τα νομίμως αλλιευμένα αλλιεύματα και ε, γίνεται μία επισήμανση με μία ετικέτα η οποία λέει πως παρανόμως έχει αλλιευθεί σε ευρωπαϊκά ύδατα και μετά έτσι κυκλοφορεί σε αγορές μας. Λοιπόν, για οποιονδήποτε κυκλοφορεί στον κλάδο αυτό πρέπει να σας πω πως όταν αποκαλύπτεται ε, πως κάποιος που κάνει κάτι τέτοιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει οι ποινές να είναι αυστηρότατες. Θέλουμε να ποινικοποιηθεί το αδίκημα γιατί μιλάμε για μια εγκληματική πράξη και θα πρέπει να χάνουν την άδεια άσκησης επαγγέλματος. Να μην έχουν το δικαίωμα να εμπορεύονται πλέον στον κλάδο της αλίας. Ξέρω ότι υπάρχει μια παράνομη διεθνής εμπορία λαθραλευμάτων. Εμείς θα πρέπει να την εκριζώσουμε να την καταστήλουμε με τον αυστηρότερο δυνατόν πρώτο και ε, συμφωνώ με τα όσα είπε η Ισαμπέλα. Χρειαζόμαστε τη διεθνή, ε, χρειαζόμαστε τη διεθνή βούληση για να εξασφαλίσουμε ότι όλα αυτά θα λειτουργήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω κι εγώ, λέει η Πρόεδρος, να κάνουμε τη σειρά μου κάποια σχόλια. Κυρίως για τα σημεία 9 και 10 της έκθεσης αυτής. Όπου κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να έχουμε μια διατύπωση η οποία θα είναι πιο κλειστή κυρίως όταν μιλάμε για τις εισαγωγές, είτε προέρχονται από ε, χώρες ε, για τις οποίες, στις οποίες έχει ε, δοθεί το σύστημα αυτό γενικευμένων προτιμήσεων, είτε γιατί πρόκειται για χώρες με τις οποίες έχουμε συμφωνίες τέτοιου είδους για την αλληλεία. Γιατί και στις δύο περιπτώσεις για να εκδοθούν τα πιστοποιητικά, τα εξαγωγικά ε, πιστοποιητικά για τις χώρες αυτές, είτε για να τους δεχθούν οι παρεκκλήσεις από τους κανόνες καταγωγής ή οι δυνατότητες προσφέρει το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων, μιλάμε πως πρόκειται για χώρες που έχουν αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις ε, ε, για την καταπολέμηση της ε, λαθραλίας. Μιλάμε για τον έλεγχο στο λιμάνι εκφόρτωσης, όπως επίσης και τα απαραίτητα παραστατικά για το αλίευμα. Άρα λοιπόν, εάν όλα αυτά δεν ε, δεν βρίσκονται διαθέσιμα, θα πρέπει το πιστοποιητικό εξαγωγής να αφαιρείται αμέσως έτσι ώστε να γνωρίζουν τα συμβαλόμενα μέρη ότι στην περίπτωση όπου δεν θα σεβαστούν αυτές τις διατάξεις είτε έχουν κάποια προνόμια λόγω της παρέκκλησης από τον κανόνα καταγωγής είτε για κάποιο άλλο λόγο, ότι οι κυρώσεις παρόλα αυτά θα είναι αυστηρότατες. Και θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι 13 πόδα νομίζω που ε, λειτουργούν ε, να δουν ποια είναι τα καυτά σημεία στα οποία θα πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω για την καταπολέμηση της λαθραλίας και να δούμε σε ποιες από αυτές τις περιοχές οι προσπάθειες δεν είναι αρκετές. Ξέρω πως στην περιοχή του Δυτικού Ειρηνικού ας πούμε, έχουμε προβλήματα στη λειτουργία και θα πρέπει να γνωρίζουμε όλες τις επιδόσεις των υπολείπων έτσι ώστε ε, να δράσουμε σε περίπτωση που υπάρχουν τέτοιου είδους περιφερειακοί οργανισμοί στους οποίους ε, πρέπει να μιλήσουμε αυστηρά. Έχουμε, για παράδειγμα, την αλία με γρηγρή. Εκεί, πολύ σωστά, και άκουσα τι είπε ο κύριος Ντέιβις, έχουμε προβλήματα που δημιουργούνται από την έλλειψη πολιτικής βούλησης, όχι μόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και εκτός. Η Επίτροπος Αλίας έχει επαναλάβει πολλές φορές πως μπορούμε να εξασφαλίσουμε ε, ε, να εξασφαλίσουμε πως όλα τα αλλιεύματα που θα εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι νόμιμα. Ότι θα έχουμε μηδενικά ε, ποσοστά λαθραλίας. δεν την πιστεύω. Δεν νομίζω πως μπορούμε να τα καταφέρουμε. Χρειάζονται και άλλες προσπάθειες και τα θέματα αυτά, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να αναφέρονται πιο συγκεκριμένα και να φανεί ότι εμεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να λύσει το πρόβλημα επιτέλους με τον καταλληλότερο τρόπο. Στο τελευταίο εκτιμώντας όπου αναφερόμαστε στην ελεύθερη πρόσβαση Νομίζω πως η μόνη αρχή ελεύθερης πρόσβασης είναι αυτή για τα ανοιχτά ύδατα. Για τις υπόλοιπες δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια διεθνής αρχή για τα όσα είπαμε για τον 17ο αιώνα, νομίζω ότι αυτά έχουν ήδη περιοριστεί και εντάξει, ελευθερία πρόσβασης, ναι. Ε, στα διεθνή ύδατα, στην ανοιχτή θάλασσα, για τίποτα ε, άλλο δεν θα πρέπει να ισχύσει. Κάτι το οποίο πρέπει να υπογραμμίσω είναι το πρόβλημα της βιοπικιλότητας που πολύ σωστά αναφέρει η συγγήτρια, η λαθραλία δημιουργεί προβλήματα κοινωνικά, οικονομικά. Έχουμε αθέμητο συναγωνισμό και προβλήματα περιβαλλοντολογικά. Και για το σημείο αυτό πιστεύω πως θα πρέπει βέβαια να τα αναφέρουμε, αλλά δεν θα πρέπει να μην δίνουμε τη δέουσα σημασία στις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις αυτής της λαθραλίας. <coughs> Θα πρέπει λοιπόν ήδη από το σημείο 1 να αναφερόμαστε στις τρεις αυτές διαστάσεις, περιβαντολογική, κοινωνική, οικονομική. Τώρα για τον νέο οργανισμό ή φορέα υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών νομίζω ότι εδώ είναι μάλλον υπερβολικά τα όσα ζητάμε. Ίσως καλύτερα θα έπρεπε εδώ να πιέσουμε στο θέμα των εμπορικών κυρώσεων που θα μπορούσαμε να επιβάλλουμε. Για τον νέο αυτό φορέα νομίζω είναι κάπως πρόημα, πρόημο να το αναφέρουμε. Ίσως αργότερα. Για το 2015 όταν λέμε μεγάλες δυνάμεις ε, να μην αναφέρουμε την Κίνα γιατί νομίζω ότι η Κίνα είναι ένα παράδειγμα προς αποφυγή στην περίπτωσή μας για τα όσα δεν πρέπει να κάνει κανείς ε, σε επίπεδο αληθικής συμπεριφοράς ή τουλάχιστον σε ε, δράση εντός των δικών τους ε, πόδα. Νομίζω πως η Κίνα δεν είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσαμε να έχουμε κατά νου. Ας μιλάμε για μεγάλες δυνάμεις και ο καθένας σας κατανοεί ποιες είναι αυτές. Σύμφωνα με την κρίση του 2021 δεν μπορώ να συμφωνήσω με το θέμα της Ιντερπόλ, αλλά είναι μια προσωπική άποψη και ενδεχομένω να έχετε κάποιους λόγους ε, ουσίας που θα μπορούσαν να με μεταπίσουν. Ωραία λοιπόν. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να κάνει και αυτή κάποια σχόλια. E η Επιτροπή θα ήθελε και αυτή να συγχαρεί την κυρία Λέβιν για την έκθεσή της που αποτελεί μια σωστή συγκεκριμένη ανάλυση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στον κόσμο της αλληλίας, της παράνομης αλληλίας δείξετε, δώσετε έμφαση σε θέματα, το θέμα όσον αφορά σε κοινωτικό επίπεδο, σε επίπεδο οργανισμών. Συμφωνούμε με την ανάλυση που κάνατε. Συμμεριζόμαστε επίση μερικέ από τι συστάσει σα. Θεωρούμε, όπω και πολλά μέλη εδώ ανέφεραν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παίξει ένα κινητήριο ρόλο σε αυτόν τον αγώνα κατά τη παράνομη αλίας. Η κυρία Δαμανάκη το έχει επαναλάβει εξάλλου ότι η στρατηγική της θα είναι μηδενική ανοχή όπου και αν γίνεται αυτή η δραστηριότητα. Αυτό το μήνυμα πρέπει να περάσουμε στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό και όπως και υπογραμμίσατε ε, η Αλία δεν γνωρίζει όρια. Θα πρέπει δηλαδή να κάνουμε τον αγώνα τόσο στα ε, χωρικά ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και έξω από αυτά. Θα πρέπει λοιπόν να συντηρήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε για τον αγώνα για την καταπολέμηση της παράνομης Αλίας, τόσο επίπεδο χωρών μελών αλλά στο επίπεδο της Επιτροπής, καλώς και των ε, υπηρεσιών που έχουν να κάνουν με τον έλεγχο αυτό. Αυτή η υπηρεσία έχει τα μέσα και ε, θα πρέπει στο μέλλον, όπως υπογράμμισε η κυρία Τρότμαν, να δει μήπως ε, αν οι χώρες μέλη έχουν τα κατάλληλα μέσα για να αποκτήσουν τη σωστή πληροφόρηση, ενημέρωση όσον αφορά την παράνομη αλληλεία και να την προωθήσουν. Να μην μείνουμε δηλαδή στο στάδιο της συλλογής πληροφοριών, θα πρέπει... Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε αυτόν τον αγώνα. Υπάρχουν πολλοί ε, που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτόν τον αγώνα. Υπάρχουν δραστηριότητες σε εθνικά επίπεδα που συμμετέχουν σε δραστηριότητες σε τρίτες χώρες για την καταπολέμηση της παράνομης αλληλείας και είναι σημαντικό να λάβουμε μέρος σε αυτή την προσπάθεια. Εμείς θα πρέπει να βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες για να αναπτύξουν μηχανισμούς ελέγχου της παράνομης αλίας. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μέσω των ε, συμφωνιών αλίας που έχουμε με αυτές τις χώρες. Επίσης, μέσω της Ευρωπαϊκού Ταμείου να μπορέσουμε να κάνουμε αξιολόγηση και να αναπτύξουμε ε, τις δυνατότητες που υπάρχουν για να μπορέσει κανείς να κάνει αυτό το έλεγχο. Διότι σε ορισμένες περιπτώσεις ορισμένοι δεν καταλαβαίνουν ότι ε, αυτή η δραστηριότητα, η παράνομη, έρχεται, ε, αποτελεί αθέμητο ανταγωνισμό, ανταγωνισμό στην παραδοσιακή αλία και είναι κατά της βιοποικιλότητας και κατά των ουσιαστικών συμφερόντων τους. Είναι επίσημα σημαντικό να πούμε ότι χρειαζόμαστε μέσα για να γίνει αξιολόγηση των ε, επιδόσεων σε παγκόσμιο επίπεδο να δούμε τις αξιολογήσεις αυτές. Επίσης να έχουμε ένα μητρό των ε, ε, αλλιευτικών πλοίων. Χαιρετίζουμε αυτή την πρόταση. Τώρα, για την εγκληματικότητα. Αυτή η δραστηριότητα, η αποτελεί ένα έγκλημα. Συμφωνούμε. Να δούμε δηλαδή το θέμα της ποινικοποίηση αυτής. θα πρέπει να ενισχυθούν οι κυρώσεις για όσους δεν κάνουν σεβασίους του κανόνες όσον αφορά τη συντήρηση των αποθεμάτων. Επίσης, και όπως είπε και η Πρόεδρος, ε, υπάρχει το θέμα της, ε, ε, του ελέγχου της όλης διαδικασίας του προϊόντος μέχρι που καταλήγει στην αγορά. Θα πρέπει να κάνουμε τα μέγιστα γι' αυτό, να έχουμε καλύτερο έλεγχο στην αγορά και εδώ η αγορά παίζει ένα σημαντικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο. Γι' αυτό θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες σε αυτό. Όντω αυτή η έκθεση, και έχω εδώ ακούσει και κάποιε προτάσει που όλα αυτά οδηγούν στην προσωστή κατεύθυνση, ε, περιμένουμε τι προτάσει και φυσικά θα επανέλθουμε με τη θέση τη Επιτροπή πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά όπω και να έχει το θέμα, η Επιτροπή ήδη χαίρεται με το διάλογο. Χρειαζόμαστε τη σύρρηξή σα για έναν αγώνα ο οποίος είναι καθημερινός. Ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν στη συζήτηση. Έχω εντυπωσιαστεί από την υποστήριξή σας που είναι τόσο ενθαρρυντική. Είναι καλό να υπάρχει συνένεση όταν επιχειρούμε κάτι. Καταρχήν ε, θα γίνει συνάντηση των σκιωδών αργότερα για να συζητήσουμε λεπτομερέστερα τις προτινόμενες τροπολογίες και προσθήκες στην έκθεση. Συμφωνώ με πάρα πολλά από αυτά που είπατε. Ε, διατυπώθηκαν και κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις από τον Chris Davis σχετικά με το πώς μετράτε η αποτελεσματικότητα. Δεν είμαι εγώ ειδικό πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά ο ΦΑΟ κάνει διαπραγματεύσεις για την επίδοση του κράτους σημαίας. Υπάρχουν επίσης διεθνείς συμφωνίες ε, όπως ε, η συμφωνία για τα ηχθή αποθέματα κλπ. Που υπάρχουν δηλαδή συμφωνίες σχετικά με το τι πρέπει να κάνει για να έχει σωστές επιδόσεις ένα κράτος. Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό και η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει ευθύνη και να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους και τις περιφερειακές και να, λειτουργήσουν στα πλαίσια περιφερειακής συνεργασίας για την εποπτεία και να δώσουν έμφαση και σε τεχνικά μέτρα παρακολούθηση σκαφών και VMS κλπ. Ε, για όλα αυτά υπάρχουν έγγραφα που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση προς τα ε, διεθνή πρότυπα. Αυτή τώρα είναι μια προσπάθεια να κάνουμε ένα βήμα ακόμη παραπέρα, γιατί ε, η καταγραφή των αλλιευμάτων είναι ένα θέμα. Θα πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο, κάτι ακόμη. Ε, μιλήσατε για τη διάσταση της αγοράς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το δούμε γιατί όλα αυτά τα ψάρια κάπου καταλήγουν. Πού καταλήγουν. Όπως είπε ο κύριος Στίβενσον, γίνονται τώρα μεταφορτώσεις στην ανοιχτή θάλασσα, αλλιεύματα ανακατεύονται με άλλα παράνομα και νόμιμα και στο τέλος όλα γίνονται νόμιμα με εισαγωγικά. Οπότε κάτι πρέπει να κάνουμε. Προτείνουμε και μια απαγόρευση των μεταφορτώσεων στην θάλασσα και το θέμα της Ίντερπολ. Κοιτάξτε, ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά παράνομα ψάρια και αυτά κάπου καταλήγουν. Άρα χρειάζονται έρευνες για να βρούμε ποια είναι τα λιμάνια, πού γίνεται η, μεταμορφ... μεταφόρτωση, πού καταλήγουν τα λιεύματα, σε ποια σούπερ μάρκετ. Γι' αυτό χρειάζονται οι αρμοδιότητες διεξαγωγής έρευνας που θα στοχεύουν ακριβώς σε αυτές τις δραστηριότητες. Γιατί αυτά είναι διακρατικά φαινόμενα. Μπορεί να είναι κάποιος Ευρωπαίος ο ιδιοκτήτης του σκάφους και να κρύβεται πίσω από μια εταιρεία η οποία έχει την έδρα της σε φορολογικό παράδεισο και ίσως το σκάφος να φέρει σημαία ευκαιρία. Το πλήρωμα μπορεί να είναι Φιλιππινέζι, ο πλήρχος μπορεί να είναι από την Νότια Αμερική και τα αλλιεύματα να αλλιεύονται έξω από την Αφρική και να καταλήγουν, να ε, εκφορτώνονται κάπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να καταλήγουν στη Σουηδία. Οπότε τι θα κάνουν. Αυτό είναι ένα μυστήριο έγκλημα και χρειάζεται σε επίπεδο αστυνομιών συνεργασία επίσης για να γίνουν σύντονες οι προσπάθειες. Τώρα, για την ερασιτεχνική αλία, την ψυχαγω... αναψυχής την αλία. Πρέπει να φροντίσουμε ώστε ό,τι γίνεται στους κόλπους της Ένωσης να είναι νόμιμο. Και δεν πρέπει να είναι πρόσχημα και κάλυψη η ερασιτεχνική αλία ή αλία αναψυχής για να γίνεται λαθραλία. Αυτό είναι απαράδεκτο. Πρέπει να φροντίσουμε και εδώ ότι η αλληλεία που διεξάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι νόμιμη. Αυτό είναι η απόλυτη βάση. Δεν μπορεί να μας πάρουν στα σοβαρά διεθνώς αν δεν είμαστε σοβαροί στα του οίκου μας και στη μικρή κλίμακα και στη μεγάλη κλίμακα. Μπορεί να υπάρχουν Ευρωπαίοι που να είναι ιδιοκτήτες σκαφών που ε, δραστηριοποιούνται στην ανοιχτή θάλασσα. Και αυτές οι περιπτώσεις πρέπει να ερευνηθούν και να επιβληθούν κυρώσεις και ποινικέ κυρώσεις, αλλά έχουμε και άλλα μέσα στη διάθεσή μας. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε εδώ το Ταμείο Αλίας, το Ευρωπαϊκό ε, Ταμείο Αλίας και να αφαιρεθούν πόροι από εκεί. Να μην έχουν ε, την οικονομική υποστήριξη από τους φορολογουμένους ε, αυτό είναι το ελάχιστο ω κύρωση που μπορούμε να προβλέψουμε. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Φράγκα, μιλήσατε για την ελεύθερη πρόσβαση. Η ανοιχτή θάλασσα είναι το 64% των ωκεανών της γης. Δεν είναι μικρό κομμάτι, είναι μεγάλο. Όταν λοιπόν ε, αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι σήμερα η επιδίνωση της ατμόσφαιρας και των ωκεανών του πλανήτη ε, είναι ραγδαία και πλήττει και αφορά όλη την ανθρωπότητα. Και όχι μόνο τη σημερινή γενιά, αλλά και τις επόμενες. Είναι οξύ το πρόβλημα και πρέπει κατεπηγόντως να το αναγνωρίσουμε. Επίσης, δεν το ανέφερα και ιδιαίτερα στην έκθεση, αλλά το 50% του διοξιδίου του άνθρακα που απορροφάται από το φυσικό οικοσύστημα, απορροφάται από τους ωκεανούς και η ικανότητα απορρόφησης του διοξιδίου του άνθρακα μειώνεται ταχύτατα. Και αυτό οφείλεται μεταξύ άλλων στην επιδείνωση των θαλασσίων οικοσυστημάτων. Και γιατί, γιατί τα, ε, ε, γιατί αλλιεύομαι ε, ψάρια τα οποία δρούν αρπακτικά στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε στα πλαίσια του παγκοσμίου οικοσυστήματος το πρόβλημα των ωκεανών που μας ανήκουν, ανήκουν σε όλους. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε ότι κάποια ε, οικονομικά συμφέροντα μικρά που δεν ε, σταματούν μπροστά σε τίποτα να δημιουργούν τέτοια μεγάλη βλάβη και σε εμά και στις επόμενες γενναίες. Γι' αυτό χρειάζεται μια, ε, ε, χρειάζονται ανεξάρτητοι φορείς αξιολόγησης που να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους, να ελέγχουν τους πόδα και να θέσουν αυτό το θέμα πολύ ψηλά στην ε, παγκόσμια ημερήσια διάταξη. Και η διεθνής κοινότητα έτσι θα μπορεί να επιβάλλει κυρώσει σε αυτούς που δεν τήρουν όλες αυτές τις συμφωνίες που εδώ και δεκαετίε υπάρχουν αλλά δεν εφαρμόζονται. Το, υπάρχει συμφωνία για τα ηχθή αποθέματα από το 1995, το άγκος από το ε, πίσω από τη δεκαετία του 1990 και δεν έγινε τίποτε σχεδόν. Τώρα είναι η ώρα να ισχυροποιήσουμε λιγάκι αυτές τις συμφωνίες και δηλαδή να τις εφαρμόζουμε, γιατί αν τις εφαρμόζαμε δεν θα υπήρχαν όλα αυτά τα προβλήματα. Αυτό είναι το ωραίο με τις συμφωνίες. Ευχαριστώ πολύ. Θα συνεχιστεί η συζήτηση αυτή στην επόμενή μας συνεδρίαση και θα έχουμε και εκπροσώπους της Κίνας, της Ιαπωνίας και των Ηνωμένων Πολιτειών στη συνάντηση αυτή για να υποβάλλετε προθεσμίες. Έχετε μέχρι τις 20 Ιουνίου. Εάν λοιπόν θέλετε να προετοιμάσετε τις τροπολογίες σας, μπορείτε να τις καταθέσετε μέχρι και τις 20 Ιουνίου. Ευχαριστούμε λοιπόν και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την κυρία Λόεβεν και θα κάνουμε την συνάντηση που είναι και κλεισμένων των θυρών, που είναι η ανταλλαγή απόψεων με εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις αλληλευτικές συμφωνίες με τρίτες χώρες και τις ανεξελίξεις διαπραγματεύσεις. Επαναλαμβάνω, επαναλαμβάνω ε, για τους συναδέλφους